Καλησπέρα σα Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Σα παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία. Καλησπέρα σας λοιπόν. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξη και θα ήθελα να σας ε, ανακοινώσω κάποιες αλλαγές. Λίγο ησυχία όμως παρακαλώ. Eh, les tengo que comunicar Να σα διαβάσω λοιπόν κάποιε αλλαγέ για να δούμε αν συμφωνείτε. Καταρχά, η κυρία Ρόντουστ ε, θα πρέπει να απουσιάσει από τις 5 και μετά και γι' αυτό ζήτησε το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη που είναι η ανταλλαγή απόψεων για την κοινή αλληλευτική πολιτική στην οποία είναι συγχύτρια να συζητηθεί μετά από το σημείο 6 ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Δαμανάκη. Η οι συγκητέ των προηγούμενων σημείων, οι κύριοι Φερέιρα και Ρωμέ Βαϊρουέδα, δέχτηκαν. Επομένως, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τους υπολείπους, ε, μπορούμε να το προχωρήσουμε έτσι. Επίσης, η κυρία Φιγκερέιντο θα αντικαταστήσει τον κύριο Φερέιρα στο σημείο υπαριθμών 7 της ημερήσιας διάταξης, διότι ο κύριος Φερέιρα απουσιάζει. Και με αυτές τις δύο αλλαγέ ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, ως τροποποιήθηκε. Επίσης να σας ανακοινώσω ότι ως συνήθως ε, η ε, συνεδρίαση μεταδίδεται στο κανάλι του Κοινοβουλίου μέσω διαδικτύου. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 26 Σεπτεμβρίου του 2011 και της 10 και 11 Οκτωβρίου 2011. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης αύριο το απόγευμα, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Ανακοινώσεις της Προέδρου, δεν υπάρχει ανακοίνωση και να περάσουμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλη η κάρτα. Καταρχάς έχουμε την έκθεση του κυρίου Ριβελίνη για δεύτερη ανάγνωση, περιοχή της Συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο. Όπως θα θυμάστε, η έκθεση του κυρίου Ριβελίνη είχε λάβει μία καταρχήν συμφωνία με το Συμβούλιο στον τριμερή διάλογο στις 22 Ιουνίου, κατόπιν οι νομικές υπηρεσίες των αρμόδιων ε, θεσμικών οργάνων συνεργάστηκαν προκειμένου να έχουμε μια οριστική διατύπωση του νομοθετικού κειμένου. Το περασμένο μήνα είχαμε και ένα σχέδιο ε, κειμένου οριστικό και τώρα μπορούμε πλέον εμείς εδώ στην Επιτροπή μας να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό σε δεύτερη ανάγνωση. Δεν ξέρω εάν ε, ε, θέλει το λόγο ο κύριος Ριβενίλη, προφανώς ε, προτείνει να εγκρίνουμε το κείμενο, τροποποίηθηκε ε, από το Συμβούλιο. Εάν δεν έχει τίποτα λοιπόν να διευκρινίσει ο κύριος Ριβελίνη, μπορούμε να ψηφίσουμε απευθείας. Ψηφίζουμε λοιπόν. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra la... Se cierra... Σε cierra la votación. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ και μία κατά. Εγκρίνεται λοιπόν το νομοθετικό ψήφισμα και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει το Δεκέμβριο. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Χάγκλουντ για την παράταση κατά ένα χρόνο της αλλιευτικής συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βασιλείου του Μαρόκου. Τη διαθέτεται, την έχουμε συζητήσει και τώρα απλώς θα πρέπει να ψηφίσουμε. Μισό λεπτό, έχουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Ο κύριος Χάγκλοντ θέλει το λόγο τώρα ή μετά. Perdón, pero yo hago lo que tengo que hacer. Eh, muy bien. Eh, en primer lugar, someto a votación las enmiendas 1 y 2 a... Λοιπόν, ψηφίζουμε τις τροπολογίες 1 και 2 στην παράγραφο 1 που είναι πανομοιότυπες. Άρχεται η ψηφοφορία. Se, cierra la votación. Πέρασε της ψηφοφορίας. Pues por 11 votos a favor y 8 en contra queda adoptada. 11 ψηφοί υπέρ, 8 κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία υπαριθμών 3 καταπίπτει, επομένως ε, άλλαξε η σημασία της ψηφοφορίας και ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra la votación. ψηφοφορίας. 12 ψήφοι υπέρ, 8 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται το κείμενο λοιπόν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Χάγκλοντ. Κύριε Χάγκλοντ, έχετε το λόγο. Ε, I just wanted to inform... Ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να σας ενημερώσω ότι αυτά που συζητήσαμε στη τελευταία συνεδρίαση ε, για το ψήφισμα δώσαμε καλέ συμβουλέ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη συμφωνία, γιατί εκπνεύσει το το Φεβρουάριο, το πρωτόκολλο μάλλον, όχι συμφωνία. Έχω εργαστεί ήδη γι' αυτό και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορους συναδέλφους. Πάντως φαίνεται δεν ικανοποιητική η συμφωνία, άσχετα τώρα με την έκβαση της ψηφοφορίας. Ε, θα έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, και με τους ε, εκπροσώπους των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα και ούτως ή άλλως θα περάσει και η έκθεση από την Ολομέλεια κάποια στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για την έκβαση της ψηφοφορίας σχετικά με την παράταση της συμφωνίας αυτής. Ε, εφ' εξής ε, θα συζητούμε το περιεχόμενο της μελλοντικής συμφωνίας με το Μαρόκο και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Πάντως, σε σχέση με την ψηφοφορία, λυπάμαι πραγματικά που ε, παρότι ήμουν σκιώδης ε, δεν συζητήσαμε τον κύριο Χάγκλουν. Τέσσερις-πέντε φορές προσπάθησα να του μιλήσω. Για λόγους που μου διαφεύγουν δεν κατέστη δυνατό να συναντηθούμε. Ε, ο κύριος Χάγκλουν προσέγγισε την πρόεδρο, καλά έκανε. Ε, αλλά όπως και για τις υπόλοιπες εκθέσεις υπάρχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ποιος ήταν, εγώ ήμουν σκιώδης. Πέντε. Πέντε φορές προσπάθησα να συναντηθώ με τον ε, κύριο Χάγκλουντ. Παρόλα αυτά εκείνος ε, ε, προσπαθούσε ταυτόχρονα να έρθει σε επαφή με την πρόεδρο. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Υπέρ φυσικά της υποβολής προφορικής ερώτησης, αλλά ήθελα να το πω αυτό. Ευχαριστώ, είναι σαφές δεν θα ήθελα να κάνουμε συζήτηση. Κύριε Χάκλουν, σας δίνω το λόγο και μετά τέρμα η συζήτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο διακεκριμένος συνάδελφός μου, ο κύριος Σέκεντεκ. λυπάμαι που ε, έχει την αίσθηση ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο. Είναι αμφίδρομη διαδικασία δυστυχώς. Ε, μετά την αρχή μας συζήτηση δεν διέκρινε την πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμβαστική σε συμβιβασμό. Πάντως για το μελλοντικό πρωτόκολλο πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επικοδομητική συζήτηση παρά τη διάσταση των απόψεων που έχουμε διαπιστώσει σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου από τις οποίες μας ψηφίσαμε. Ελπίζω να συνεχίσουμε για το ψήφισμα, να εργαζόμαστε με επικοδομητικό ε, τρόπο. Χαίρομαι που ο κύριος Καντέκ ε, είναι υπέρ του, της ιδέας του ψηφίσματος. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να δημιουργούμε προς ε, τριβές και διενέξει εκεί που δεν υπάρχει ένας λόγος. esta cuestión. Καλώς. Ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Μαρία Δαμανάκη. Η Επίτροπος όμως δεν είναι παρούσα ακόμα. Είναι καθοδόν μας είπανε. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους δεν πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα ε, να αποχωρήσουν από την αίθουσα προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και κλεισμένων των θυρών.